Colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to make a start because we have... Συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε διότι στις 4 και 4 έχουμε ψηφοφορία και θέλω να προλάβουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν, μια και βρίσκονται εδώ τα βασικά μας μέλη, ε, να ξεκινήσουμε. Σημείο 1. Έκριση της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ σημειώστε ότι το σημείο 9, η ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή θα πραγματοποιηθεί πριν το σημείο 5 και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται η ημέρησια διάταξη. Σημείο 2. Ε, η, ε, το γλωσσικό καθεστώς δεν έχουμε διερμηνία ε, από τα κροατικά και γοηδελικά. Ε, ε, το, ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, οπότε παρακαλώ να έχετε μαζί σας τις κάρτες σας. Προχωράμε στο σημείο 3. θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγή για του σκοπού κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτο διεθνού προστασία. Η εισηγήτριά μα είναι η Σιλβή Γκυγιό με 95. Τροπολογίε έχουν υποβληθεί και συνάδελφοι όπω γνωρίζετε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό ε, κατάλογο. Ε, Στόχο τη πρόταση τη Κομισιόν είναι να ε, θεσπιστεί ένα τέτοιο κοινό κατάλογο δίνω το λόγο στην εισηγήτρια και θα δώσω μετά το λόγο σε όποιους ευρωβουλευτές θέλουν να πάρουν το λόγο. Σίλβη, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν πλέον παρά μόνο 94 τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να υποφεληθώ από την παρουσία κάποιων από τους σκιώδεις Θέλω να ευχαριστήσω και τους απόντες ε, για τη βοήθειά τους και γιατί τελικά η αντίληψη την οποία θέλησα να προτείνω φαίνεται ότι ακολουθείται από τους περισσότερους ε, από τους σκιώδεις και νομίζω ότι μέχρι τώρα ε, τα πράγματα εξελίχθηκαν θετικά. Σε μια δεύτερη φάση θα μπορέσουμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες να θυμίσω ότι η αντίληψη την οποία προτείνω την ακολουθεί και το Συμβούλιο. Γιατί αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε για τις λεγόμενες ε, ασφαλείς χώρες και η υπηρεσία αυτή ξεκάθαρα επιφορτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στον συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, πέρα από τις χώρες οι οποίες είναι σε ξεχωριστό, αν θέλετε, σε ξεχωριστή ομάδα, υπάρχουν ε, πέντε βασικά θέματα. Καταρχάς, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεύτερον, διαδικασία αναθεώρησης της λίστας για προσθήκη και αφαίρεση. Τρίτος τομέας, διαδικασία διακοπής της συμμετοχής της χώρας εφόσον υπάρξει χειροτέρευση ευνίδια της κατάστασης, τέταρτον μεθοδολογία και πέμπτον θεμελιώδη δικαιώματα. Πρώτη ομάδα, η σύνδεση ανάμεσα στους εθνικούς καταλόγους και τον ευρωπαϊκό κατάλογο. Υπό ΚΑΠΑ όλοι οι σκιώδεις συμφωνούν με την ενισχυμένη συνεργασία οι προθεσμίες οι οποίες προτείνονται μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά υπάρχει πάντως η επιθυμία σαφής να ενταχθούμε σε μια διαδικασία εναρμόνισης. Μου φαίνεται δυνατό να προτίσουμε μια λύση έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα των εθνικών καταλόγων και να προωθήσουμε ένα ουσιαστικό κατάλογο ευρωπαϊκό. Αυτά προβλέπονται όλα να γίνουν σε λογικές προθεσμίες και στα πλαίσια αυτής της μεταβατικής φάσης ελπίζω να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια μεταβατική λύση. Είναι ένα θετικό σημείο θα έλεγα αυτό ε, για την διαδικασία. Το δεύτερο θέμα αφορά την διαδικασία αναθεώρησης προσθήκης μάλλον χωρών. Ε, εδώ έχουν κάποιοι σκιώδεις προσθέσει ε, κάποιες τρόπους για να λάβουμε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτό. Αυτό νομίζω είναι χρήσιμο γιατί θα μας επιτρέψει να προετοιμάσουμε τη μεταβατική περίοδο. Και αυτό θα έλεγα αφορά και στο θέμα στο οποίο ανάφερα προηγουμένως. Το τρίτο θέμα είναι η διαδικασία διακοπής συμμετοχής αν υπάρξει ευνίδια χειροτέρευση της κατάστασης σε μια χώρα που θεωρείται ασφαλής. Κάποιοι σκιώδεις ε, θέλησαν να ενισχυθεί η δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης, γρήγορης προσαρμογής της ευνίδιας αλλαγής. Από την άλλη θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει ένας μηχανισμός διακοπής ε, πιο ευέλικτος ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις έγκαιρα. Πρέπει να είμαστε και στις δύο περιπτώσεις, όχι οι γραφειοκράτες, αλλά να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα. Ευέλικτοι, αλλά και σαφείς, γιατί αν η διαδικασία δεν είναι σαφής, τότε θα δημιουργηθεί μια κάποια αβεβαιότητα. Και αυτό θα θίξει και τις ίδιες τις χώρες, όπως όμως και την του συγκεκριμένου οι οποίοι θέτουν το συγκεκριμένο ερώτημα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Εδώ υπάρχει συμφωνία γενικότερα για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων οι οποίοι φύγονται από τη διαδικασία αυτή. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ε, την αποδοχή των προτάσεων της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα πλαίσια των ετοιμάτων που είχαμε εκφράσει στο παρελθόν. Πέμπτο σημείο η μεθοδολογία. Έχουν δοθεί χρήσιμες διευκρινήσεις, λίγες τροπολογίες κατετέθησαν μετά από τις προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε νομίζω ότι στηρίζουν οι σκιώδεις τις προτάσεις τις οποίες εγώ κάνω στο επίπεδο μεθοδολογίας. Είπαμε ότι η μεθοδολογία είναι καθοριστικού, έχει καθοριστικό ρόλο και διαπιστώσαμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προτείνει μια μεθοδολογία ξεκάθαρη προς το παρόν. Συνεπώς θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Η ύπατη αρμοστία άλλωστε έχει καταλήξει σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Θέλω να είμαι σαφής στην φάση αυτή, όπως ελπίζω ότι ήμουν και στο παρελθόν στις απαντήσεις που έδωσα προς τους σκιώδεις. Εμείς ε, δεν πρόκειται να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σύνολο βιομηχανικής επεξεργασίας ευρωπαϊκού επίπεδου όλων αυτών των θεμάτων. Αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι μια λειτουργική ευρωπαϊκή λίστα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και λίγο καιρό θα πρέπει να δώσει στο Γραφείο Ασύλου την δυνατότητα να συλλέγει σωστά τις πληροφορίες για να φέρει πέρα στην εντολή του. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς εδώ, να προβλέψουμε μια διαδικασία διαβούλευσης και το εννοώ ε, που να περιλαμβάνει και ανεξάρτητες, ε, ανεξάρτητα μέλη γιατί τώρα πλέον το Γραφείο Ασύλου θα έχει νέες αρμοδιότητες. Εδώ η πατιαρμοστία μας είπε ότι καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα με μας. Λοιπόν, ε, δεν θα φτιάξουμε κάτι το περίπλοκο, θέλουμε κάτι το λειτουργικό και απλό. Και δεν θα πρέπει, θα έλεγα, να αγνοήσουμε τις ρήτρε προστασίας σε σχέση με ε, το ε, νέο σύστημα. Το θέμα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα τώρα ε, φανταστήκαμε, αλλά νομίζω ότι η Βρετανική πλευρά σαν παράδειγμα μας δείχνει εδώ το δρόμο και έχει λειτουργήσει το σύστημα και η Γαλλία έχει στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που έκανε πρόσφατα πάρει μέτρα που θα ήταν χρήσιμα να τα εξετάσουμε. Η επόμενη συνάντηση των σκιωδών θα γίνει στις 7 Ιουνίου μετά από τη συζήτηση σήμερα. Θα, συζητήσουμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις και ελπίζω ότι οι αποφάσεις μας θα μας επιτρέψουν να κλείσουμε τη διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν, να ψηφίσουμε δηλαδή ε, λίγο πριν από το τέλος του μήνα για να συνεχίσουμε την εξέταση του κειμένου αυτού που αξίζει το ενδιαφέρον μας και να μην χρησιμοποιηθεί το κείμενο αυτό για λόγους οι οποίοι θα έλεγα είναι διαφορετικοί από τους βασικούς του στόχους. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά στις ομιλίες σας. Όσοι πάρετε το λόγο από τώρα να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Γκυλιόμ. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Έδειξε υπομονή. Εγώ δεν θα είχα αυτή την υπομονή και ήταν και ιδιαίτερα ευγενής και κομψή στη μεθοδολογική της αντιμετώπιση. Να σας παρουσιάσω τη θέση μου με λίγα λόγια για τις τροπολογίες τις οποίες έχουμε καταθέσει. Εγώ θα συμφωνήσω πλήρως με την διευκρίνηση των διαφορών ανάμεσα στους εθνικούς καταλόγους και στους, στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Αν φύγει μια ασφαλής χώρα από τον ευρωπαϊκό κατάλογο δεν μπορεί να παραμείνει στον εθνικό γιατί τότε θα έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια ε, χωρίς λόγο δωρεάν. Λοιπόν, ε, δεν θα είναι άμεσα συγκεκριμένος ο κατάλογος ο ευρωπαϊκός, θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρξουν συγχύσεις, επικαλύψεις ε, και θα δημιουργηθεί επίσης και σύγχυση στην ακολουθητέα πρακτική έτσι ώστε να επιλέγουμε σωστά τις αιτήσει χορήγησης ασύλου. Πρέπει να περάσουμε μακροπρόθεσμα σε μια ενιαία ευρωπαϊκή λίστα ασφαλών χωρών θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τον τρόπο προσθήκης των χωρών αυτών, γιατί αλλιώς θα χάνουμε την ώρα μας. Η διαδικασία την οποία κάνουμε σήμερα θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται αν θέλουμε να προσθέσουμε μια τρίτη χώρα. Ε, για την κοινή λίστα δεν θα είναι αποτελεσματική παρά μόνο αν συνοδεύεται από συμφωνίες επανεισδοχής Νομίζω ότι αν έχουμε κάποιες ασφαλείς χώρες αλλά οι χώρες προέλευσης δεν δέχονται ε, την α, επανεισδοχή τότε δεν έχει νόημα. Εγώ προσθέτω επίσης ε, και το θέμα ε, των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ευρωπαϊκής βοήθειας. Δεν αρκεί μόνο ένα σύστημα κυρώσεων, πρέπει να δίνει κίνητρα για την επανεισδοχή. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχω να κάνω σε επίπεδο πολιτικής ομάδας. Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή ήταν καλυμμένα αλλά είναι περίπλοκη μέχρι τώρα. Πάντως πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα και νομίζω ότι έχουμε ένα σημείο συμφωνίας έτσι ώστε να καταστεί το μέσο αυτό πραγματικά αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη. Αλλιώς θα έχουμε πάντα τις ίδιες δυσκολίες με όλα τα δράματα γιατί την ώρα που, που, που δουλεύουμε η τραγωδία συνεχίζεται. Είδαμε τι συνέβη στην Μεσόγειο αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω κάτι άλλο de l'ensemble, du contenu de l'ensemble des amendements que nous avons déposés. Alors, je vous remercie. Thank you very much. Uh, the ECR shadow is Mr. Halafako, please. Thank you, Chairman. Σκιώδης των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, κύριε Χάλα Άχο. Η ECR, η ομάδα μου, πιστεύει ότι για να είναι αποτελεσματικό ο κατάλογος πρέπει να είναι φιλόδοξος και να μην είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και να μπορεί να αντιδρά ταχύτατα σε αλλαγές στις καταστάσεις σε τρίτες χώρες. Παρόλο που καταρχήν προτιμούμε ένα ενιαίο κατάλογο στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένω ένα τέτοιο κατάλογος να αποδειχθεί λιγότερο εύκαμπτο από τον εθνικό ή του εθνικού κατάλογους. Γι' αυτό έχουμε κάποιε επιφυλάξει σχετικά με την τροπολογία 47, σύμφωνα με την οποία χώρε οι οποίε θεωρούνται μη ασφαλεί από την Ένωση θα διαγράφονται και από του Εθνικού καταλόγου. Θα πρέπει λοιπόν ο κατάλογο τη Ένωση να είναι το ίδιο εύκαμπτο και φιλόδοξο όπω και αυτό των χωρών μελών για να προσφέρει προστιθέμενη αξία και ιδίω εάν πρόκειται τελικά να αντικαταστήσει του εθνικού. Συμφωνούμε επίση με την τροπολογία 69 σύμφωνα με την οποία κάθε χώρα που έχει καθεστώτος υποψήφιας χώρας θα πρέπει να θεωρείται ασφαλής και να διαγραφεί από τον κατάλογο. Αν μια χώρα δεν είναι ασφαλής, δεν θα πρέπει να είναι υποψήφια για ένταξη. Όπως είπα πριν, δεν είναι απόλυτα σαφές τι σημαίνει η επιταχυμένη διαδικασία για ετούντες άσυλο που έρχονται από ασφαλή χώρα. Είναι όμως κρίσιμο αυτό για να έχει αποτέλεσμα και αξία ο προτινόμενος κατάλογος. Ας αρκεστώ σε αυτά για την ώρα. Ο Γιος Άλμπρεχτ των Πρασίνων. Ευχαριστώ στα αγγλικά θα σχολιάσω στην βάση των όσων μου έχει σημειώσει ο Τζιν Λάμπερτ που είναι ο δικός μας ε, εισηγητής. Εμείς προτείνουμε πρώτα την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν, διότι θεωρούμε ότι η έγκρισή της θα θέσει σε κίνδυνο την αρχή της α, κατά περίπτωση εξέτασης κάθε υποθέσεως ασύλου. Δεύτερο, όμως, εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να διατηρήσει την πρόταση, εμείς έχουμε καταθέσει ορισμένες τροπολογίες που θεωρούμε ότι αποσαφηνίζουν ορισμένα πράγματα και συμπληρώνουν το έργο της εισηγητρίας. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να είναι μερική εντολή, να εξετάσει δηλαδή τις αρχές που έχουν σχέση με κάθε ε, χώρα μέλος ξεχωριστά. Με κάθε χώρα ξεχωριστά. πρέπει να είναι εγγυημένα τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα για όλους. Προτείνουμε επίσης τροπολογίες για να διαγραφούν παραπομπές στις διαγραφές χωρών για να μειωθούν οι αιτήσει ασύλου. Επίσης, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε συγκεκριμένη προθεσμία για την κατάργηση των εθνικών καταλογών, διότι δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα χρειαστεί η επανεξέταση για να δοθούν οι σχετικές κατευθύνσεις με χώρες προελεύσεως κλπ. Συμφωνούμε επίσης ότι οποιαδήποτε χώρα διαγράφεται από τον κατάλογο της Ένωσης θα πρέπει να διαγράφεται και από, τον κατάλογο, τους κατάλογους μάλλον των ε, χωρών τους εθνικούς καταλόγους δηλαδή. Αυτό θα πρέπει να είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία και αν μια χώρα διαγραφεί επί μια διετία θα πρέπει το αποτέλεσμα να είναι σαφές και η χώρα αυτή να μην θεωρείται πλέον ασφαλής. Σημειώστε επίσης ότι θα επαναφέρουμε τις τροπολογίες μας 34, 35 και 109. Ευχαριστώ. Λεμπερτών και Φερών για το ENF. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εμεί καταθέσει μία τροπολογία γενικής απορρίψεως, διότι θεωρούμε ότι είναι απολύτως αποτυχημένη η πολιτική ασύλου για την ώρα. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, θεωρούμε ότι πρέπει να πάυσουν απολύτως οι διαπραγματεύσεις για ένταξη της χώρας αυτή στην Ένωση, γιατί η Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η χώρα αυτή αντιμετωπίζει σημαντικότατες δυσκολίες και παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, ιδίως ό,τι αφορά ε, τους τζιχαντιστές που ε, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης και το Κόσοβο είναι μια διαφθαρμένη χώρα όπου απαλήφονται οι ε, χριστιανικές μειονότητες. εκθέσεις όπως ε, αυτή που έχουμε μπροστά μας υποσκάπτουν την κυριαρχία των μελών και των χωρών δηλαδή και μας βρίσκουν απολύτως αντίθετους. Τέλος, ο κύριος Κύρκος παρακαλώ. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική προσέγγιση της εισηγήτριας ε, και χαίρομαι που πρώτα προσεγγίζουμε τη μεθοδολογία, απεμπλέκουμε τον κατάλογο των χωρών από τη διαδικασία έγκριση, αναθεώρηση, εναρμόνιση κτλ. Και στην ουσία αφήνουμε το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με την μέθοδο που είναι το πιο σημαντικό και να μην εμπλακεί με την επιλογή των κρατών που εκεί οι πιέσει είναι πολύ μεγάλε από και από την επικαιρότητα. Εμεί στην Ελλάδα περάσαμε με το πακέτο τη συμφωνία, περάσαμε και την έγκριση τη Τουρκία ω ασφαλή χώρα ε, με μια συζήτηση που κράτησε δύο ώρες. Φυσικά δεν ήταν σε βάθος. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπόκειται σε πίεση του Κοινοβούλου για λόγους ε, της επικαιρότητα. Άρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από αυτό το ξεχωριστό και περιμένουμε φυσικά την απάντηση της μελέτης της ΕΑ για να συζητήσουμε το ουσιαστικό που είναι η ένταξη της κάθε μίας χώρας. Ευχαριστώ. Thank you. And uh, Mrs. on of uh, Martina Anderson. Η κυρία Βεργίου, που εκπροσωπεί την Μαρτίνα Άντερσον. Ευχαριστώ και Πρόεδρε, καθυστέρησα λίγο, όμως δεν ήθελα να εξεταστεί το κείμενο χωρίς θέση της πολιτικής μας ομάδας, γιατί είναι απούσα η σκέφτη συγκεκριά μας που είναι η κυρία Άντερσον και η οποία έχει συνεργαστεί καλά με την κυρία Γκυλιόμ, όπως και η Πράσινη, και εμείς καταρχήν απορρίπτουμε το σύνολο της προτάσεως της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε μάλιστα ότι εν ώψη της εξελίξεως ε, τι καταστάσεω σε ορισμένε χώρε. μέλη πρέπει να φτιαχτεί μια λίστα μη ασφαλών χωρών και οι προφορίε που λαμβάνουμε το λιγότερο που μπορεί να πει κανεί είναι ότι οι χώρε που ενδέχεται να περιληφθούν στον κατάλογο των ασφαλών χωρών, τουλάχιστον το μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτέ τι χώρε. Και μάλιστα σημαντικά, διότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτέ τι χώρε που όχι μόνο δεν μπορούν να υποβάλουν έτσι ασύλου, αλλά που δολοφονούνται. Αυτά πάντα έχουμε υπόψη όταν προχωρούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και είμαι απόλυτα κα, ε, κατάπληκτη όταν βλέπω ότι είναι τον, τρο, τον δρόμο παίρνει η κατάσταση. Πρόκειται για όχι δράμα απλώς ασύλου, δράμα προσφύγων και τελικώς θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών στην Μεσόγειο. Αυτό δείχνουν οι στατιστικές. 3.700 σχεδόν νεκροί στην Μεσόγειο, 2.000 από την αρχή του χρόνου. Αν κάνει κανείς την προβολή θα φτάσει 7-8.000 μέχρι τέλους του έτους. Πόσο θα συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι με τόσο θανατηφόρα αποτελέσματα. Και κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ε, σταθούν υπόλογες απέναντι στην ιστορία και με τρώτα λόγια μου. Σας ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην ε, ΛΥΠΕ. Ε, θα έχουμε και τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν ξέρω αν η κυρία Γκυγιόμ θέλει να πει κάτι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Σιλβί. Προσβλέπουμε στην ε, συνέχιση των εργασιών. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 4, αγαπητοί συνάδελφοι θα παρακαλούσα τον ε, Διευθυντή και την ε, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ε, Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να έρθουν στο βήμα. Μέχρι να έρθουν ο κύριος Οφλάχερτη και η κυρία Ζάιτεν Στίκερ, να σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Έχουμε τη χαρά σήμερα να καλωσορίσουμε εδώ σήμερα τον κύριο Οφλάχερτη, τον νέο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την κυρία Φράουκε Ζάιτεν Στίκερ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα μα παρουσιάσουν την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα του 2016. Η έκθεση συνοψίζει και αναλύει σημαντικέ εξελίξει όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Διαπιστώνει τι πρώτο έχει σημειωθεί και τι ε, εμπόδια συνεχίζουν να υπάρχουν και ε, αναλύει τα βασικά θέματα που ε, διέπουν τη συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την άξη των τριμερών διαλόγων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Σάιτενστικερ και μετά τον κύριο Φλάχερτη. Πρώτη φορά προεδρεύω σε συνεδρίαση που βρίσκεστε εσεί εδώ. Νομίζω θα ακούσουμε πρώτα την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Φλάχερτη. Σας καλωσορίζω θερμά και τους δύο. Κυρία Ζάιντεν Στίκερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που μας προσκάλεσατε εδώ να σας παρουσιάσουμε την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ε, εκτίμησή μας για τις συνεχείς προσπάθειές σας να συμπεριλαμβάνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και σας ευχαριστώ και για την συνεργασία σας. Ήταν μεγάλη μας χαρά που συναντήσαμε κάποιους από εσά στον οργανισμό μας την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, κάθε χρόνο προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ετήσια έκθεση για να γίνει πιο εύχρηστη και να είναι και πάντα επίκαιρη για τις συζητήσεις περί πολιτικής ε, που ε, πραγματοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί κάθε κράτος μέλος έχει δικές του προτεραιότητες ε, και δικές του προκλήσεις. Θα προσέξατε ότι έχει αλλάξει ο τίτλος της έκθεσης, τώρα λέγεται «Έκθεση θεμελιωδών δικαιωμάτων» και και τώρα πια αναφέρουμε το έτος δημοσίευσης και όχι τα έτη που καλύπτει η έκθεση. Με έμφαση στο παρόν έτος θέλουμε να δείξουμε ότι είναι επίκαιρη η έκθεση αυτή σε αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική. Τα δεδομένα που δημοσιεύουμε στην έκθεση στις περισσότερες περιπτώσεις αναλύονται ε, από την προοπτική των θεμελιωδών δικαιωμάτων και παρουσιάζονται ε, υπό συγκρίσιμη μορφή για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, αυξάνουμε και τον αριθμό και τη σημασία που δίνουμε στις νομοδοτήσεις στην έκθεση. Αφενός τις δημοσιεύουμε ξεχωριστά σε όλες τις ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε έτσι να γίνουν πιο εύχριστες ε, και χρήσιμες και για εσάς και τους συναδέλφους σας ε, και εδώ στις Βρυξέλλες και στις πατρίδες σας για να λυθούν υπόψη τα στοιχεία αυτά κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών. Οι γνωμοδοτήσεις ε, συμπληρώνουν τις νομικές γνωμοδοτήσεις για την προγραμματισμένη νομοθεσία που ετοιμάζουμε κατόπιν εντολής ε, των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από τις νομοδοτήσεις αυτές εκπονούνται κατόπιν εντολής της δικής σας επιτροπής, ε, για παράδειγμα όσον αφορά τον ε, κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης σε ένα θέμα που μόλις συζητήσατε. Άλλη γνωμοδότηση ήταν για τους δείκτες θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της έκθεσης πρωτοβουλίας σας για το, την εγκαθίδρυση μηχανισμού ε, για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εμπειρογνωμοσύνη μας με τον τρόπο αυτόν, διότι έτσι διασφαλίζουμε ε, τη, να εξετάζονται πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την νομοθετική διαδικασία. Ε, τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης ε, δεσπόζουν στο θεματολόγιο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό για το Διοικητικό Συμβούλιο και για τον οργανισμό μας στο σύνολό του να εκπονήσουμε εκθέσεις και οι γνωμοδοτήσεις αυτές καλύπτουν το θεμελιώδες δικαιώμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, ε, την ε, εισαγωγή ε, μέτρων νόμης μετανάστευσης για να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων και την σημασία της ένταξης των μεταναστών. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί σωστά το μεταναστευτικό, ε, σεβόμενη πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στι εργασίε του οργανισμού μας ε, και σε πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα και βραχυπρόθεσμα. Για να μπορέσουμε όμως να πετύχουμε κάποιες αλλαγές, χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο δυναμικό ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι περιφερειακός παράγοντας, πρέπει να βρίσκεται στον κέντρο των συζητήσεων. Η μεταναστευτική πολιτική είναι η πολιτική που μεταβάλλεται πιο γρήγορα αυτή τη στιγμή εντός Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό για να υπάρχει βιωσιμότητα και αξιοπιστία όσον αφορά τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να παίξουν σημαντικό ρόλο τα θεμελιώδη δικαιώματα και κατά το σχεδιασμό νέων πολιτικών και κατά την ε, εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, θα πρέπει να υπερασπιστεί την αρχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο στο θέμα αυτό. Του Λεχθέντος θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, διευθυντή μας, τον κύριο Οφλάχερτη, ο οποίος θα σας παρουσιάσει κάποια ε, σημεία κλειδιά της έκθεσης πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, συνάδελφοι, θα συμφωνήσω με την Πρόεδρό μου, ευχαριστώντας σας για την πρόσκληση και υποδοχή και την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την ετήσια έκθεση. Ξέρετε ότι γίνεται αποδεκτή από τη Διαχειριστική Επιτροπή μετά από τις προτάσεις της διοίκησης της υπηρεσίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην Βιέννη για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκαναν μέχρι σήμερα. Αγαπητά μέλη, το 2015 και θα είμαι ειλικρινή ήταν μια κακή χρονιά. Υπήρξε η παναχώρηση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμένων. Υπήρξε αύξηση της ανεξέλεκτης ρητορική που προκαλεί προβλήματα στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις συνδεόμενες αξίες. Αν διαβάσετε, όταν διαβάσετε τα κεφάλαια της έκθεσής μας θα το δείτε αυτό. Θα ήθελα να θέσω ένα πλαίσιο απλά. Το πρώτο πλαίσιο, όπως είπε η Πρόεδρος, αφορά στα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου. Δεν θα σας δώσω περαιτέρω στατιστικές τις οποίες γνωρίζετε καλά. Αλλά κάθε φορά που αναφερόμεθα στην κρίση αυτή, έχουμε να κάνουμε με μια κρίση αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως προς αυτό λοιπόν εκτιμούμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή σας έχει παρακολουθήσει από κοντά την εξελισσόμενη κατάσταση και σας ευχαριστούμε που συνεχίσετε να, σέφετε, να στρέφετε την προσοχή σας μέσω πολλαπλών διαδοχικών ακροάσεων στην κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όσο προχωράμε συνάδελφοι θα δείτε πολλά στοιχεία σημαντικά και λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση δείτε σαν παράδειγμα αποδείξεις ότι το 2015 υπήρξαν υπαναχωρήσεις σε πολλές χώρες που θα οδηγήσουν ή σε, οδήγησαν σε καταστάσεις επαναπροώθησης. Υπήρξαν επίσης αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι αιτήσει, κάτι το οποίο τις αιτήσει, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει επανειλημμένα σε μορφές επαναπροώθησης μη επιθυμητές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να στραφώ τώρα σε ένα, νέο, σε ένα δεύτερο θέμα, τα δικαιώματα των παιδιών. Εδώ η μετανάστευση επιβάλλεται. Ανάμεσα στο 30 και το 40% των μεταναστών είναι παιδιά. Το ποσοστό των μεταναστών που χάνουν τη ζωή τους δυστυχώς αντιπροσωπεύει 30% παιδιών. 30% ε, αυτών που πνίγηκαν στη Μεσόγειο σημαίνει ότι από το Σεπτέμβριο του 2015 δύο παιδιά πνίγονται καθημερινά και φυσικά να μην αναφερθώ στους τεράστιους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πορείας μετανάστευσης. Αν δείτε την ετήσια έκθεση, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια κάποια βελτίωση. Σε μια πρώτη φάση απαιτείται να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εντάσσοντας τις πολιτικές προστασίας της παιδικής ηλικίας, τις διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Θα πρέπει επίσης να είμαστε ταχύτεροι σε σχέση με την απονομή κυδαιμονίας για τα ασυνόδευτα παιδιά. Ο τρίτος τομέας στον οποίο θα αναφερθώ είναι η έλλειψη ανοχής και ο ρατσισμός. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάρα του 2015. Από πολλές χώρες έχουμε πάρα πολλά συμβάντα όπως επιθέσεις αντισημετικού τύπου, αντιισλαμικού τύπου, αντιτσιγκανικού τύπου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε το εύρος και το βάρος των επιθέσεων στις μειονότητες. Οι μειονότητες δεν είναι το πρόβλημα, είναι τα θύματα. Είναι ανεπαρκείς οι νομικές ρυθμίσεις ή δεν εφαρμόζονται σωστά και εν μέρη οι ρυθμίσεις αυτές. Όπως παρατηρεί η ετήσια έκθεση, οι περισσότερες από τις χώρες μας πρέπει να είναι πιο αποδοτικές στην καταγραφή και την δίωξη δίωξη των εγκλημάτων μίσους. Τώρα να μιλήσω λίγο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει μια μόνιμη προσπάθεια εξισορρόπησης της εθνικής ασφάλειας από τη μία με τα θεμελιώδη δικαιώματα από την άλλη. Η έκθεση αντικατοπτρίζει την συνεχιζόμενη σημασία και βάρος των προτάσεων περιορισμού των δικαιωμάτων επί τη βάση τριών βασικών αρχών. Νομιμότητα, αναγκαιότητα, αναλογικότητα. Εξετάσαμε τα θέματα αυτά σε βάθος κατά τη διάρκεια του 2015 μετά από αίτημα που λάβαμε από την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή για μια γνωμοδότηση για την παρακολούθηση ε, και τα θεμελιώδη δικαιώματα και καταθέσαμε την, μας, την έκθεσή μας πριν μερικούς μήνες. Να αναφερθώ σε δύο περίεργα ευρήματα. Σε πάρα πολλές χώρες υπάρχει μαζική παρακολούθηση από αυτές μόνο πέντε έχουν νομικό πλαίσιο για αυτού του είδους την παρακολούθηση. Δεύτερον, υπάρχει μια πολλαπλότητα συστημάτων εποπτείας και επίβλεψης στα διάφορα κράτη-μέλη. Στα πλαίσια αυτής της πολλαπλότητας υπάρχουν θέματα ανεπαρκούς επαϊωσύνης και ανεπαρκών αρμοδιοτήτων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. Κλείνοντας αγαπητά μέλη, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να μου επιτρέψετε να κάνω τέσσερις προτάσεις. Πρώτον, θα θέλαμε να ζητήσουμε την προσοχή σας για τις 41 συστάσεις τις οποίες περιλαμβάνει η έκθεσή μας. Είναι σταθμισμένες και νομίζω ότι είναι όλες ευφυείς σε εισαγωγικά το λέω αυτό, αλλά θα σας βοηθήσουν να κάνετε σωστές ενέργειες σε εθνικό επίπεδο και καλύπτουν όλες τις θεματολογικές ε, πλευρές με τις οποίες ασχολούνται. Δεύτερον, η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι η καρδιά της λήψης νομοθετικών αποφάσεων. Εδώ εσείς παίζετε ένα σημαντικό ρόλο, αλλά δεν συμβαίνει δυστυχώς σε όλους τους τομείς αυτό. Τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να είναι υπαρκτά παντού πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα, σαν παράδειγμα με πιο ξεκάθαρο τρόπο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τρίτον, θα πρέπει να ισχύσουμε την, ενισχύσουμε την κατάρτιση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να διευρύνουμε τα προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες μέλη ε, να είναι προγράμματα τα οποία να έχουν την απαιτούμενη οικονομική κάλυψη και να έχουν πάντα σαν βασική βασικό χαρακτηριστικό τον σεβασμό της χάρτας των θεμελιωδών. Προχωρώντας λοιπόν, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι δική σας, είναι το ανεξάρτητο κέντρο θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και αριστείας κοινοτικής στον τομέα αυτό. Ε, δίδει εξαιρετικά δεδομένα σε αιτήσια βάση, χρησιμοποιήστε τα αυτά, χρησιμοποιήστε τις νομικές βάσεις, χρησιμοποιήστε τις νομοδοτήσεις και τις συστάσεις, έτσι ώστε ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο στα όργανά μας και στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, εμείς στην υπηρεσία μας είμαστε στην διάθεσή σας σε καιρούς δύσκολους. Um, σας ευχαριστώ και τους δύο που μιλήσατε με σύντομο τρόπο. Είναι όντως λεπτομερέστατη η εκθεσή σας, είπατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε όμως και κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να ακούσετε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών και να τον κλείσουμε εφόσον συμφωνείτε. Εσείς επίσης ζητήσατε, είναι. Θα διαβάσω λοιπόν τα ονόματα και θα κλείσουμε τον κατάλογο. Έτσι λοιπόν, τα εξή ονόματα. Πεςτε τώρα όμως αν θέλετε να μιλήσετε κι εσείς. Άρα όλοι, λίγο πολύ. Δύο λεπτά λοιπόν. Εδώ κλείνει ο κατάλογος. Εάν έρθει κι άλλος τώρα, υποστηρίξτε με, δεν θα δώσουμε το λόγο σε άλλον η άλλοι, παρακαλώ, τηρήστε το όριο των δύο λεπτών. Γνωρίζετε ότι έχουμε και ψηφοφορίες μετά. Ο Μπόνι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την έκθεση που τη βρίσκω πολύ χρήσιμη και σημαντική. Είναι καλά δομημένη, έχει και ας πούμε ήπιες συστάσεις soft recommendations, γιατί είναι εκφρασμένες πιο πολύ σαν γνωμοδοτήσεις της, του οργανισμού σας, σε μια προσπάθεια στήριξης των χωρών μελών, στις πολιτικές που ασκούν. Θα ήθελα να έρθω σε δύο θέματα. Αφενός προστασία δεδομένων και κοινωνία της ε, πληροφορικής και των πληροφοριών, είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι κανόνες αυτοί, δηλαδή αναγκαιότητα, νομιμότητα και αναλογικότητα. Στη δική μου χώρα, στη σχετική νομοθεσία για τις αστυνομικές δυνάμεις και μαζική επιτήρηση και αντιτρομοκρατία, δεν υπάρχει κατάλογος σοβαρών εγκλημάτων, δεν υπάρχει δικαστικός έλεγχος εκ των προτέρων, πράγματα τα οποία βρίσκω προβληματικά, δηλαδή προβλήματα διαχείρισης και ελέγχου αυτών των δραστηριοτήτων. Δεν το λέω επειδή δεν μου αρέσει η χώρα μου, τη λατρεύω τη χώρα μου. Αλλά κάπου διαγνώσκω μια τάση, μια, μια ένταση αν θέλετε, ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ελευθερία. Χρειάζεται λοιπόν να αναλύσουμε τις συστάσεις σας, να τις κάνουμε και πιο διαφανείς για τους πολίτες. Στην Πολωνία, που είναι η χώρα που λατρεύω, έχουμε τώρα και οργανωμένους πολίτες που ζητούν νομοθεσία για την τρομοκρατία. Τώρα να προσθέσω κάτι για αυτά που λέτε για ρατσισμό, ξενοφοβία και έλλειψη ανοχής. Συμφωνώ με το πρώτο μέρος της ε, παραγράφου αυτής της εκθέσεώς σας σε σχέση με κάποιες δραστηριότητες και κάποιες πολιτικές. Δυστυχώς στη χώρα μου η κυβέρνηση αποφάσισε να διαλύσει το Συμβούλιο που ήλεγχε τις δραστηριότητες κατά της ξενοφοβίας κλπ. Και που αποτελείται από πολλούς εκπροσώπους πολλών οργανισμών και τους έδινε τη δυνατότητα να δράσουν όλοι μαζί. Ευχαριστώ κύριε Βεργιά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω ξεκινώντας να ευχαριστήσω εκ νέου τους εκπροσώπους της υπηρεσίας η επάρκεια και η ακρίβεια της παρουσίασης της έκθεσής τους ε, μου άρεσε. Μου άρεσαν επίσης τα σημεία προσοχής τα οποία προωθούνται φέτος και τα οποία δείχνουν ακριβώς και την ικανότητα επιλογής της σειράς την οποία έχει η υπηρεσία. Είπατε ότι το 2015 ήταν μια κακή χρονιά, πήγαν πίσω τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπήρξε μια κρίση των δικαιωμάτων και των αξιών. Πολλοί είμαστε σε αυτήν την Επιτροπή που θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Ίσως όχι τόσο στο πρώτο σημείο, ένα σημείο επί το οποίο θα ήθελα να επιμείνω, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου σε διάφορες χώρες στα πλαίσια των πολιτικών μετανάστευσης στο θέμα της μη επαναπροώθησης και των ομαδικών ε, εκδόσεων Νομίζω ότι υπάρχει και θέμα για την προστασία αυτών που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες και πρόσφυγες, για το θέμα των παιδιών όλο και περισσότερα. Πολλά παιδιά χάνουν όλο και περισσότερα τη ζωή τους στη θάλασσα, πολλά παιδιά χάνονται στην πορεία τους Είχα πάει στην Ιταλία πριν 15 μέρες και μπορέσαμε να δούμε ακριβώς τον μεγάλο αριθμό των παιδιών των ασυνόδευτων στις τελευταίες αφήξεις. Να πω επίσης ότι η πολιτική μου ομάδα θα επανέλθει στο θέμα αυτό και μάλιστα το βλέπουμε να περιλαμβάνεται, μην ανησυχείτε πρόεδρε θα σταματήσω εδώ, χαίρομαι που το βλέπω στο πλαίσιο της έκθεσής μας, αυτό είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί ιδιαίτερος. Η Γκουε λοιπόν θα ζητήσει κατά τη διάρκεια της επομένης συνεδριάσεως των συντονιστών να υπάρξει μια γνωμοδότηση για την κατάσταση των δικαιωμάτων των μεταναστών στα hot spot στην Ιταλία και κυρίως στην Ελλάδα για τις κρατήσεις, την διάρκεια κράτησης και την κράτηση ανηλίκων. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να διαμορφώσουμε μια εικόνα. Ε, να πω επίσης ότι πήρα μέρος στην απονομή του βραβείου Σαχάροφ, τη συνάντηση των βαβερμένων με το βραβείο Σαχάροφ. Είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. Δυστυχώς μόνο αυτό δεν κάνουμε. Ευχαριστώ. Είμαι υποχρεωμένος να σας ειδοποιώ όταν, μετά την πάροδο των δύο λεπτών. Κύριε Κίρκοπ, συγχαρητήρια στους συγγραφείς τις εκθέσεις που είναι πραγματικά ενδελεχείς. Έρχομαι στα θέματα των παιδιών κυρίως. Και πρώτα για την παιδική φτώχεια. Πολύ χαίρομαι που μπορέσαμε να φτάσουμε σε κάποιο συμβασμό μεταξύ εκείνων που θεωρούσαν ότι ε, μόνο υλικά στοιχεία έχουν κάποια ρόλο να παίξουν. Και το θεματικό. Τώρα θα ήθελα επίσης να πω για την ειδική μεταχείριση των παιδιών στα νομικά συστήματα που αναφέρεστε στο εγγραφό σας. Με ενδιαφέρει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά τυχαίνουν ειδική μεταχείριση και σε ό,τι αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες και ακόμα πιο ειδικά τις ψυχιατρικές υπηρεσίες που νομίζω δεν αναφέρονται καθόλου εδώ και που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ στην προστασία των παιδιών απέναντι σε εγκλήματα που ε, διεξάγονται μέσω του διαδικτύου. Και για τους παρόχους υπηρεσιών, εγώ ε, ήμουν στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας που μετέβη στις Ενωμένες Πολιτείες και συναντήθηκε εκεί με παρόχους υπηρεσιών γνωρίζουν τις ευθύνες τους, πάντως είναι σημαντικό να συνεχίσει να διεξάγεται διάλογος μεταξύ ημών και αυτών. Τέλος, για την ριζοσπαστικοποίηση. Όλους μας απασχολεί πολύ αυτή η ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Καμιά φορά οφείλεται στις κοινωνικές συνθήκες, καμιά φορά σε οικογενειακές. Έχουν πάντως σχέση και με την έκθεσή τους στα μέσα, κοινωνικά μέσα δικτύωσης κλπ. Και, και το διαδίκτυο. Σε ποιο βαθμό Γνωρίζω ότι αναφέρεστε στο θέμα αυτό στην έκθεσή σας, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται αρκετά πράγματα. Ως οργάνωση τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να ενθαρρύνετε δράσεις που θα αναλάβουν με τη σειρά τους οι εθνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Δυστυχώς, ε, είπα από πριν ότι είναι κλειστός ο κατάλογος πλέον. Βεβαίως το θέμα είναι τέτοιο που όποιος εισέρχεται στην αίθουσα και αντιλαμβάνεται περί πρόκειται θέλει να τοποθετηθεί. Ε, ο επόμενος, η επόμενη συνάδελφος. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές και θα ήθελα να κάνω σχόλια σε τρία σύντομα θέματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σεβασμό της προσωπικής τους ελευθερίας μόνο και μόνο γιατί είναι μετανάστες ή ε, ζητούν άσυλο υπάρχουν ε, πάνω από χίλιους ανήλικες, ανήλικους συγγνώμη, οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση αυτή. Θυμίζω ότι πέρυσι δημοσιεύθηκε μία μελέτη για εναλλακτικές λύσεις για τις διάφορες μορφές ε, κράτησης. Από τότε χειροτέρευσε η κατάσταση ε, τα κέντρα γίνονται ολοένα και περισσότερο κλειστά. Νομίζω ότι περιμένουμε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο δεύτερος τομέας είναι η συμφωνία με την Τουρκία. Έχουμε αμφιβολίες για την ομιμότητα της ίδιας της συμφωνίας. Έχουν ε, υπάρξει θα έλεγα πολλές παρατηρήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα είναι αν η υπηρεσία σας έχει αναλύσει τη συμφωνία αυτή και τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Εμείς στην ΚΟΕ στείλαμε μια αντιπροσωπεία στην Τουρκία και αυτά τα οποία είδαμε είναι ότι υπάρχει μια συστηματική παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υποχρεωτικές μετακινήσεις, πυροβολή αστυνομία στα σύνορα τους μετανάστες και θα θέλαμε να μάθουμε αν εσείς θα προετοιμάσετε μια κάποια έκθεση για την πλευρά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την παραβίασή τους και πώς θα διαμαρτυρηθείτε για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Και ο τελευταίος τομέας είναι για το νέο σώμα, το οποίο θα αντικαταστήσει την υπηρεσία Frontex και την οποία θα ψηφίσουμε σήμερα. Είναι το πρότυπο της Ευρώπης ε, φρούριο, της Ευρώπης οχυρό, που δεν θέλαμε υποτίθεται. Ε, θα έχει ε, ιδιαίτερα δικούς της τρόπους ε, χρηματοδότησης και αυτό θα την καταστήσει ακόμα πιο αδιαφανή από τη Frontex. Δεν θα βοηθήσει τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Είναι σαφής η ερώτησή σας, αλλά πρέπει να επιμείνουμε να τηρείτε τον χρόνο ομιλίας. Πίτερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση και να θέσω μια ερώτηση. Η γενική παρατήρηση είναι ότι το κράτος δικαίου, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι προϊόντα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τι γίνεται λοιπόν με τα κράτη-μέλη που θέλουν, δεν θέλουμε τέτοια δημοκρατία, Θέλουμε δημοκρατίες μη φιλελεύθερες. Ε, έτσι λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα επανακαθοριστούν. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε αυτές τις χώρες. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τη στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι την περιγράφεται. Υπάρχουν διάφοροι διάφορες μορφές ε, διάκρισης, ε, υπάρχει ε, ο διαχωρισμός κατά την εκπαίδευση. Νομίζω όμως ότι το το χειρότερο είναι η καταναγκαστική μεταγκατάσταση Ρωμά σε κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορείτε να κάνετε, πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε να σταματήσουμε τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τζούρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Είπατε ότι υπάρχουν πράξεις μυσαλλοδοξίας στην Ευρώπη. Αυτό που με ανησύχησε ήταν ότι παραλείψατε τη μυσαλλοδοξία εις βάρος χριστιανών μεταναστών, διότι είδαμε πράξεις βίας σε κέντρα μεταναστών ε, ή ε, στις ε, στις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι μετανάστες. Ε, για παράδειγμα, ε, μία μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρθηκε σε τέτοια περιστατικά πριν δύο περίπου εβδομάδες και επίσης ε, τέτοιες πράξεις συνοδεύονται συνήθως από πράξεις που αποτελούν καταφανή παραβίαση του κράτους δικαίου και παραλείπουν οι αρχές ε, να ενημερώσουν το κοινό και να αναλάβουν δράση. Έχω επίσης ε, μία ερώτηση. Δεδομένων των τραγωδιών που βλέπουμε κατά την ε, παράνομη μετανάστευση, ακούσαμε ότι πνίγηκαν εκατοντάδες άνθρωποι τις τελευταίες μέρες. Αυτοί λοιπόν που κερδοσκοπούν σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να ε, διωχθούν και να τους πάμε στα δικαστήρια, διότι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για οργανωμένο κίνημα και οι ανθρώπινες αυτές τραγωδίες ε, είναι ευθύνες κάποιων που κερδίζουν από αυτές. Ε, η κυρία Ινετφέλντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία παρατήρηση περισσότερο παρά ερώτηση. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, για τις ακούραστες προσπάθειές του ε, στην, ε, πρόθεση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαβάζοντας την έκθεση αυτή και τις προηγούμενες, βλέπω ότι αναλύουμε πολύ σωστά τι πάει στραβά και καταχωρίζουμε τις ε, παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ε, τα διαπιστώνω όλα αυτά με αυξανόμενη δυσαρέσκεια, διότι τι κάνουμε για όλα αυτά. Στην Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή εκπονούμε προτάσεις για έναν μηχανισμό για την διατήρηση της δημοκρατίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διασφάλιση του κράτους δικαίου. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν ο οργανισμός ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να παίξει ρόλο όχι μόνο στην ε, διαπίστωση των παραβιάσεων των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά αν μπορεί να βοηθήσει και ε, στην εξάλληψη των ε, προβλημάτων, ε, διότι δεν είναι απλά αντικειμενικοί λόγοι, συχνά υπάρχουν πολιτικοί λόγοι και έλλειψη πολιτικής βούλησης για αντιμετώπιση των θεμάτων. Δεν παραβιάζονται κατά λάθο τα ανθρώπινα δικαιώματα, πάντα κάτι τέτοιο αποτελεί το αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν στις αναλύσεις σας και στις συστάσεις σας θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερη προσοχή στο πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερη πολιτική υποστήριξη για την καταπολέμηση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Βαλέρο, σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση σχετικά με μία ομάδα που δεν αναφέρεται εδώ στην έκθεση τους ε, ανθρώπους ε, χωρίς, ε, χωρίς χαρτιά, χωρίς έγγραφα. Στους απάτριδες. μπορεί να υπάρχει εντολή απέλασης, η οποία όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Τώρα με τη νέα πολιτική μετανάστευσης που υποδεχόμαστε πολλούς από χώρες εμπόλεμες. Προσπαθούμε να ε, στείλουμε πίσω όσους ε, έχουν απορριφθεί οι αιτήσει τους. Ε, αναρωτιέμαι τώρα και πόσοι κρύβονται στις χώρες μας, στη Σουηδία, την πατρίδα μου για παράδειγμα. μιλάμε για τους ε, απάτριδες, ανθρώπους χωρίς έγγραφα. Ε, εάν λοιπόν απορριφθεί η αίτησή τους, ε, κρύβονται πολύ απλά. Ε, δεν μιλάμε για τους, τους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε με τα δικαιώματά τους στις χώρες μας. Και όχι μόνο αυτούς των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί, να εκτελεστεί, αλλά και αυτούς που ήταν ενδεχομένως με προσωρινή άδεια παραμονής, έχουν μείνει για πολλά χρόνια, έχουν ενταχθεί πολύ καλά ε, αλλά τώρα με την άφηξη τόσων νέων ε, δεν τους χορηγείται τελικά μόνιμη άδεια παρομενής, ε, αλλά επιστρέφονται αναγκαστικά. Υπάρχει και εδώ κίνδυνος να κρύβονται οι άνθρωποι αυτοί αντί να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις ομάδες αυτές ε, που ε, κινδυνεύουν ε, να καταλήξουν χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να κρύβονται τελικά στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λοριστίν, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την προηγούμενη ερώτηση, διότι τώρα συζητάμε για το σύστημα του Δουβλίνου και βλέπουμε ότι και την ε, ανανέωσή του ή την ε, μεταρρύθμισή του. Βλέπουμε λοιπόν ε, δευτερογενείς μετακινήσεις. Ποια είναι λοιπόν η θέση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την ελευθερία, με την ελεύθερη κινητικότητα, αυτό που συνδέεται με την οικογενειακή επανένωση, και τέτοια θέματα, διότι βλέπουμε από τη μία ότι στη Σουηδία και άλλες χώρες ε, η ελεύθερη κινητικότητα δημιουργεί προβλήματα. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, πώς θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ πλήρη και ενδιαφέρουσα έκθεσή σας. Περιέχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Tack Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ για την έκθεση. Στο κεφάλαιο 4 αναφέρεστε στην ένταξη των Ρωμά. Συμφωνώ με τι γνωμοδοτήσει που παρουσιάσατε. Θα ήθελα ωστόσο να θέσω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των Ρωμά. Ζούμε σε εποχές ε, όπου η πολιτική και η κοινή γνώμη ε, δημιουργούν αντιθέσεις ε, μεταξύ διαφόρων ομάδων. Βλέπουμε πολλά λαϊκιστικά κόμματα, αλλά ακόμα και αξιοπρεπή εντός εισαγωγικών κομμάτων. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε να δοθεί περισσότερη προτεραιότητα στα θέματα των Ρωμά στο πολιτικό θεματολόγιο. Η κατάσταση για 6 εκατομμύρια ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι πρέπει να φύγουν από τις χώρες τους ε, λόγω ε, σημαντικών διακρίσεων, δίωξης, φτώχειας και για άλλους λόγους. Πολλοί από αυτού ε, που ε, χρησιμοποιούν λοιπόν τη δυνατότητα τη ελεύθερη κινητικότητα ε, τελικά αντιμετωπίζουν μεταχείριση χειρότερη από σκυλιά. Οι άνθρωποι που φύγανε από τις χώρες τους κατά τον πόλεμο των Βαλκανίων κινδυνεύουν να σταλούν πίσω σε εντός εισαγωγικών ασφαλείς χώρες είναι ασφαλής για τους υπολείπους, όχι όμως για τους Ρωμά. Επίσης, τι γίνεται με τους απάτριδες, ποιος προστατεύει τα δικαιώματά τους, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ και εδώ έχουμε πολλούς Ρωμά λόγω του πολέμου των Βαλκανίων και του καθορισμού των συνόρων. Υπάρχουν ε, λοιπόν πολλά θέματα τα οποία πρέπει ε, να, ε, στα οποία πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο πολιτικό μας θεματολόγιο. Ευχαριστώ. Η Σιλβή Ιβόν Κάουφμαν είναι η τελευταία ομιλήτρια. Ένα λεπτό αν μπορείτε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς καθυστέρησε η πτήση μου και δεν μπόρεσα να είμαι εδώ εγκαίρως. πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για την έκθεσή σας. Έχετε στην σελίδα 22 ένα τμήμα της έκθεσής σας όπου μιλάτε για την Eurodac. Ε, λέτε ότι έχετε μοιράσει ερωτηματολόγια στα κράτη-μέλη. Και λέτε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και να γίνεται δακτυλοσκόπηση τους. Ε, θα ήθελα Λοιπόν, να ρωτήσω στο ένα λεπτό. Έχετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα τρία σημεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον γραμματέα της υπηρεσίας. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τέσσερις και τέταρτο πρέπει να τελειώσουμε. Θα κάνω ό,τι μπορώ να είμαι σύντομος, λέει ο κ. Σοφλάρτη και η κυρία και θα κλείσει με τις δικές της παρατηρήσεις σχετικά με την ερώτηση την οποία έκανε ο κ. Μπόνι. Δεν, να, δεν μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες σαν χώρα, αλλά θα ήθελα να τον ενημερώσω και τα μέλη της Επιτροπής ότι θα παράγουμε στο μέλλον μια, θα έλεγα, έκθεση για την εξέλιξη των παρακολουθήσεων και τον σεβασμό των νομικών πλαισίων. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον νομίζω για όλους. Για την κυρία Βερζά έθεσε πολλά θέματα για τα θέματα των μεταναστών, τα οποία έθεσαν και πολλά άλλα μέλη της Επιτροπής. Να πω εξ αρχής ότι η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συμφωνεί ότι έχουμε να κάνουμε με μια κρίση θεμελιωδών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικότερα. Εμπλέκονται όλοι εδώ και πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλοι και σε σχέση με την Ελλάδα, όπου στην Ελλάδα έχουμε, αν θέλετε, την πρώτη προσωρινή αποστολή πεδίου στηρίζοντας τις ΜΚΟ που λειτουργούν εκεί. Το θέμα είναι ε, για τις ε, νομοδοτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, στα hot spots. Δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς ε, μέσω της έκθεσης αυτής ε, να βοηθήσουμε. Αν το πιστεύετε θα σας θα ανταποκριθούμε. Τέθηκε το θέμα και των, της ψυχολογικής στήριξης. Θα δείτε ότι για το 16 έχουμε προχωρήσει σε ειδικέ παρατηρήσεις, συστάσεις για την υγεία των μεταναστών. Και εδώ τίθεται και το θέμα της ψυχολογικής υγείας σχετικά με τους κινδύνους ε, για τα παιδιά online, του διαδικτυακούς κινδύνους, να πω ότι οι απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πεδίο προστασίας εδώ μπορεί να βοηθήσει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και στο φόρουμ που θα διεξαρθεί στις επόμενες εβδομάδες για την παρέμβαση της κυρίας Άλμπιολ. Τι κάνουμε εκεί όπου υπάρχουν κρατήσεις ανθρώπων, εμείς επισκεπτόμεθα τακτικά τα ελληνικά νησιά. Έχουμε μία μικρή ομάδα που έχει έδρα την Ελλάδα. Δίδουμε συμβουλές και συστάσεις προς τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ έτσι ώστε να αποφεύγονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό θα συνεχιστεί να γίνει σε συνεργασία με τη Frontex με την οποία έχουμε μια εξαιρετική θα έλεγα μορφή ε, συνεργασίας. Ε, έχουν τεθεί πολλά θέματα από πλευρά σας ε, που δεν απαντώνται σύντομα. Να πω πάντως ότι εμείς ε, εκεί που απειλούνται τα δικαιώματα στις αναδιόμενες λεγόμενες δημοκρατίες αλλά και στις χώρες μας παραπέμπουμε στις υποχρεώσεις οι οποίες δεν αλλάζουν και που περιλαμβάνονται στη συνθήκη. Νίντε Μίλα πάλι για και κυρία Πόστο για τα δικαιώματα των Ρωμά. Να πω ότι η υπηρεσία μας έχει καταλάβει το πρόβλημα. Η κατάσταση των Ρωμά είναι ένα σκάνδαλο για την Ευρώπη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια του χώρου ε, αμμοδιοτήτων μας για να οθήσουμε προς τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κοινοτήτων Ρωμά όπου και αν βρίσκονται και αναφέρομαι εδώ όχι μόνο στους Ρωμά αλλά και όλες τις ε, περιπλανόμενες κοινότητες για τις διώξεις εις βάρος των χριστιανικών μειονοτήτων. Ανεξαρτήτως της ε, θρησκευτική ομάδας, το ενδιαφέρον μας είναι δεδομένο εφόσον η εντολή μας τους καλύπτει. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιούρεκ ότι απαιτούνται επίσης ε, και λύσεις σε ποινικό επίπεδο για τους σωματεμπόρους δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται οι σωματέμποροι με τους μετανάστες. Η κυρία Ιντβελτ έθεσε πάρα πολλά θέματα. Να απαντήσω στην πρόσκλησή της για το πώς θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια που να οδηγούν στις παραβιάσεις που είναι καρπός πολιτικής πολύ συχνά είναι καρπός πολιτικής. Είναι συχνά επίσης και καρπός άγνοιας, έλλειψης ευαισθησίας, έλλειψης κατανόησης και έλλειψης πόρων. Πρέπει λοιπόν όλες αυτές τις διαστάσεις να τις υπογραμμίσουμε και με τα περιορισμένα μας μέσα να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε. Ε, είναι δύσκολο για μια έκθεση ε, να προλάβει κάποια γεγονότα. Είναι δύσκολο να φτιάξουν μια έκθεση για κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Ε, κύριε Φαλέρο, για τους, ε, για τους μετανάστες, τους απάτριδες και αυτούς που δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι είναι πολύ περίπλοκος ο τομέας αυτός και ο καθορισμός του μέλλοντος κάθε μετανάστη θα πρέπει να εξατομικεύεται. Δεν μπορεί να υπάρχει ομαδική απάντηση, ε, ακόμα και για τους Ρωμά. Ε, η ατομική περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η Λοριστίν για το Δουβλίνο και την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Και αυτός είναι περίπλοκος τομέας. Εδώ θα μπορέσουμε να δώσουμε μια επίσημη γνωμοδότηση προς το Κοινοβούλιο εφόσον μας τη ζητήσετε. Και τέλος, η κυρία Κάουφμαν για το Eurodac. Ίσως δεν σας κατάλαβα καλά, αλλά θα είμαι ιδιαίτερα ε, ευτυχής να τα συζητήσω τα θέματα αυτά αδίμερος. Σας ευχαριστώ αγαπητά μέλη. Η κυρία Ζάιντεν Στίκερ. Σας ευχαριστώ έλεγα πολύ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις που μας υποβάλατε, είτε πρόκειται για δικαιώματα των Ρωμά, είτε των παιδιών, είτε των χριστιανικών μειονοτήτων, για παράδειγμα. Θα συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε γύρω από τις ερωτήσεις αυτές και το ε, Διοικητικό Συμβούλιο θα μεταφέρει τις συζητήσεις αυτές που διεξάγονται εδώ στις δικές μας. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν να ε, στοχαζόμαστε για τα θέματα αυτά. Η εφαρμοσιμότητα και η δυνατότητα πρόσβασης στις ε, προτάσεις μας. Εμείς προσπαθούμε να φτάσουν οι προτάσεις μας αυτές σε διάφορα επίπεδα ε, λήψεως πολιτικών αποφάσεων. Τέλος, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε σχετικά με την πολιτική βούληση. Βεβαίως δεν μπορούμε να αυτοπεριοριστούμε, δηλαδή ε, να περιοριστούμε μονάχα στο να καταδεικνύουμε πού βρίσκονται οι παραβιάσεις. Εμείς δείχνουμε στο βιβλίο μας, στην έκθεσή μας και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές. Είναι ένα πρώτο βήμα. Συμφωνώ όμως ότι χρειαζόμαστε συζητήσεις που να στραφούν γύρω από τις πολιτικές. Η διάσκεψη που θύμισε ο ε, πρόεδρός μας, ο διευθυντής μας, το φόρουμ δηλαδή που θα ε, διοργανωθεί, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί, είστε ασφαλώς όλες και όλοι προσκεκλημένοι για να συμμετάσχετε στις συζητήσεις. Ευχαριστώ και τους δυο σας, ευχαριστώ βέβαια και το προσωπικό του οργανισμού σας που συνέταξε αυτή την πολύ ουσιαστική έκθεση. Χάρηκα πολύ για αυτά που είπατε κύριε Φλάχερτη σχετικά με το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του FRA. Και θα συστήσω σε όλους τους συναδέλφους μου να διαβάσουν ε, προσεκτικά την εκθέσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην συζήτηση. Εάν έχετε έτοιμες τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, θα αρχίσουμε στις 4 και 15 τις ε, ψηφοφορίες. Θα είδατε ήδη ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των ψηφοφοριών. Θα ήθελα να μην ξεπεράσουμε τις 6 και 15. Να είστε έτοιμοι, λοιπόν και Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προτείνω οι συντονιστές να φροντίσουν να είναι παρόντα όλα τους τα μέλη και όλοι να έχουν τις κάρτες τους για τις ψηφοφορίες. Μπορείτε παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσετε. Παρακαλώ καθίστε. Έχουμε μια πολύπλοκη ψηφοφορία μπροστά μας. Εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε προβληματάκι να μου το πείτε αμέσως. Συνάδελφοι, το σημείο 9 της ημερησίας διάταξης, πρόταξη κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, ε, που ανακαλεί τον κανονισμό 2007-2004 και τον κανονισμό 863-2007 καθώς ε, και την ε, απόφαση του Συμβουλίου 2005-267. Εισηγητής Artis Πάμπριξ, τροπολογία 103. Παρακαλώ ψηφίστε. Δεν λειτουργεί. Ε, παρακαλώ ξαναδοκιμάστε, διότι και το δικό μου δεν λειτουργήσε την πρώτη φορά. Επαναλαμβάνω. Τροπολογία 103. Μπορείτε ακόμα να ψηφίσετε. Ε, να περιμένουμε ένας ευρωβουλευτής προσπαθεί ακόμα να ψηφίσει. Δεν λειτουργεί. Ωραία, μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε αν είναι θετική ή αρνητική ψήφος σας. Μπορείτε να ψηφίσετε με το χέρι. Ένας από τους S&D λοιπόν ε, ε, ψηφίζει για να Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 102. Αρχή τη ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104, αρχή της ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη. 104 και 263 μαζί. Από κοινού. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, ε συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. εγκρίνεται οριζόντια τροπολογία 2 της Επιτροπής Μεταφορών Αρχή της Ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 122 Λογική Σκέψη 5 Αρχή της Ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 208. Αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 220. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 5, παράγραφος 1, τροπολογία 317, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 794, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 1, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός για το άρθρο 2, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 249 και 253 από κοινού. Αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 250, 251, 252 από κοινού αρχή της ψηφοφορίας. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 του εισηγητή. Αρχή της ψηφοφορίας. closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 260. Αρχή της ψηφοφορίας. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 261. Αρχή της ψηφοφορίας. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 3. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβιβασμός για το άρθρο 4. Συγγνώμη, τροπολογία 275, αρχή της ψηφοφορίας. The Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία το άρθρο 4, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 286, αρχή της ψηφοφορίας. λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 5, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 340, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 342, αρχή της ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 του εισηγητή. Αρχή της ψηφοφορία. Closed. Λήξη της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 6. Αρχή της ψηφοφορία. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 6α νέο. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 7. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 374. Αρχή της ψηφοφορίας. 374. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 395. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 405. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 406, συγγνώμη, ΑΦΕΤ 32, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 416, 417 και 418 unblock, λέει ο πρόεδρος. Όχι, 416 και 417 από κοινού, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 418, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 9, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 10, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 427, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 448 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 458 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 11. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 474. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 12. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 13. Ε, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ε, χωρίς το and third countries, αρχή της ψηφοφορίας και τρίτες χώρες. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 561. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 14. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 15, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 592, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 596, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 16. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 601. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 17. Αρχή της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 607. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 612. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 617 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίφτεται. 627 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 18, ε, το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Ακόμα μπορείτε να ψηφίσετε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική του άρθρου 19, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 6.94, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 43. Του εισηγητή. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 698. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 696. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 697 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 699 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 700. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 701. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 702. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 703 αρχή της ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 704 αρχή της ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 706 αρχή της ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 4 της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 707 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία. αρχή της ψηφοφορίας της Μόνικα Χόλμα για προφορική τροπολογία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πέντε της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 24. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική του άρθρου 25. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 726 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 26, το πρώτο τμήμα. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 7.47 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική του άρθρου 27 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 756 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 757 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική του άρθρου 28 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 29. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 30. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 32. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 33. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 807. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 34. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 35. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 8.33. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 8.35 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8.39 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική το άρθρο 36 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 861 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 862 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική του άρθρου 37 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 8.65 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική του άρθρου 38 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 41, διορθώνει ο Πρόεδρος, συμβαστική του άρθρου 39, αρχή της ψηφοφορίας, άρθρο 39. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 41, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προπολογή 883, όχι, λάθος, έχει αποσυρθεί. 896, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική των άρθρων 44-45, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική των άρθρων 46 και 49. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9-18. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 920. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9.21 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική του άρθρου 51 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική το άρθρου 52, το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της, ε, της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβαστική του άρθρου 53, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 960. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 967 και 978 όχι, 967 και άφετ 69 είναι όμοιες αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 976 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. 978 και 979 είναι ταυτόσιμες αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική του άρθρου 54 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 994 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9.95 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9.96 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. εννέα της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Αρχή τη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. 9.99. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική του άρθρου 60. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική του άρθρου 61. Αρχή της ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αφέτ 76. Αρχή της ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 1024. Αρχή της ψηφοφορίας. Closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1020. Αρχή της ψηφοφορίας. Closed. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Συμβιβαστική στο 63 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 1027 ε, ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική στο άρθρο 67 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική στο άρθρο 68 ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική στο άρθρο 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή Συμβιβαστική στο άρθρο 70. Ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 1084 ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 1087 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 10.90 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική στο 71 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στο 72 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 11.39. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 11.40. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 11.55. Ψηφίζεται. Τέλος. απερίφη. Συμβιβαστική στο 74. Ψηφίζεται. Στο 74 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Λοιπόν ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 1162 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική στα 75 με 78 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 79 με 82 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 105 ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 106 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική στην αιτιολογική 2 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 113 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 118 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 116 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 117 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική στην αιτιολογική 5 ψηφίζεται. Τέλος. 124 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 125 ψηφίζεται. Τέλος. Συμβιβαστική στην 7 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 132 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική στην εννέα, Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 138. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 139 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 140 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 142 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 143 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 144 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 146 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 145, α, συγγνώμη συναδελφοί, πηγαίνουμε στην 149, ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. Συμβιβαστική στο 14 ψηφίζετε. Τέλος. Δεκτή συμβιβαστική στην 15 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή συμβιβαστική στις 16 και 16 νέα ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή συμβιβαστική στην 17 ψηφίζεται. Τέλος Δεκτή. Στην 18 ψηφίζεται. Τέλος. Συμβιβαστική στην 20 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Στην 21 ψηφίζεται. Τέλος.

απερίφθη στη συμβιβαστική στην 22 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 196 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική στην 23 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 24. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 25. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 209 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Αλληλεία 4 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Αλληλεία 5 δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στον καθένα, λέμε πες πέντε. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 28 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 28 νέα α και 28 νέα β και την 29. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτές. 221 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική στην αιτιολογική 30 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 31 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 33 ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Προϋπολογισμός 2. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. 229 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική στην 39 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε στο τροποποιημένο κείμενο. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτό 40 υπέρ 10 κατά 5 αποχές η ψηφοφορία για την απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της ΛΥΜΠΕ ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. 44 υπέρ, 9 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Πάμπεξ. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία colleagues, uh, Αγαπητές και αγαπητοί, αντέχετε ακόμη, αντέχετε να συνεχίσουμε. Αισθάνεστε Ρωμαλαίοι και Ρωμαλαίες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για λογαριασμό της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την Post-Electoral Revision του Δημοσιονομικού πλαισίου, πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Η συγγέντρια είναι η κυρία Άτζια. Τροπολογία 1. Αν με συγχωρείτε, φαίνεται πω δεν είναι όλοι έτοιμοι ακόμη. Συμβιβαστική. Συμβιβαστική τροπολογία 1, λέει ο πρόεδρο. Αν και θα δώσω λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσει να καθίσει το άλλο. Μην λησμονείτε ότι είμαστε ακόμα σε ψηφοφορία. Καθίσατε παρακαλώ όλες και όλοι. Ωραία. Συμβαστική 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται αυτή. Τροπολογία 7. Αρχίζει. Πρόκειται για ονομαστική ψηφοφορία. Ή πάντως ηλεκτρονική. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 17 τροπολογία αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτή. Υπαριθμόν 18 αρχίζει. Τέλος. εγκρίνεται. Συμβαστική 3 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 27 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 28 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Στο σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ, 4 κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ακολουθεί η επόμενη ψηφοφορία, ανταλλαγή πληροφοριών Ακολουθεί λοιπόν η ψηφοφορία για την έκθεση, για την οδηγία, για την ανταλλαγή πληροφοριών για επικόους τρίτων χωρών όσον αφορά το σύστημα έκρης ποινικών μητρώων. Ρωτώ πρώτα αν ο εισηγητής επιθυμεί να λάβει το λόγο. Όχι, έχει καλώς. Τότε λοιπόν σημειώστε ή μάλλον να ρωτήσουμε τον εισηγητή. Έχουμε έτοιμα από το Λαϊκό Κόμμα για την ονομαστική ψηφοφορία για ορισμένες τροπολογίες αρχής γινωμένης από την 8 υποστηρίζετε την αίτηση αυτή του Λαϊκού Κόμματος. Ο εισηγητής την ε, δέχεται. Το ίδιο ονομαστική ψηφοφορία από τους πράσινους για 36, 45, 50 και 52. Μάλιστα θετική γνώμη και αυτή. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Αρχίζουμε με την συμβιβαστική 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8α. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ωραία. Έληξε και αυτή. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8β σε τμήματα. Πρώτο, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Άρα, προχωρούμε στην τροπολογία 36. Ονομαστική ψηφοφορία προπολογία 36. 36. Διότι, μάλλον λόγω του αποτελέσματος της φοβορίας που μόλις έγινε. Πηγαίνουμε στην 36. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Αρχίζει. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, ξεχάστε αυτή την ψηφοφορία. 37 και 38, ταυτόσιμες. 37 και 38, ταυτόσιμες. Αρχίζει η ψηφοφορία και για τις δύο. Πέρας. Εγκρίνονται. 14. 14 και 41 ταυτόσημες. 14 και 41. Ταυτόχρονα λοιπόν ψήφος. Πέρας. Εγκρίνονται. 43 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται ή εγκρίνεται 44 αρχίζει πέρας εγκρίνεται 46 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 47 αυτή η κυκλοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 49 αρχίζει. έκανα ένα λάθος. Έχει εκπέσει 49, δεν θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Διαγράφουμε την ψηφοφορία και πηγαίνουμε στην υπαριθμόν 50. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 52. Άρχεται. Ονομαστική πάλι. Τροπολογία 52. Πέρας. Εγκρίνεται. 53. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 54. Αρχίζει. Ονομαστική. Τέλος. Εγκρίνεται. 55. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ονομαστική. Τέλος. Εγκρίνεται. 16. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτή. 17 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 57 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Τροπολογία 19 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 58-59 είναι ταυτόσιμες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 9 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τα εκτιμώντας. Ένα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Αρχίζει η ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Αρχίζει η ψήφος. Δεν ψηφίζουμε τη συμβαστική 4 διότι, διότι εγκρίθηκε η 36. Άρα, έδειξε η ψήφος για την 26 και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Συμβαστική 5 πρώτο τμήμα. Αρχίζει η ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Αρχίζει ψήφος. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Αρχίζει η ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 45 πέντε ψήφοι υπέρ, δύο κατά και τέσσερις αποχές. Τώρα αρχίζει η ψήφος παρενομαστική για την χορήγηση της διαπραγματευτικής εντολής. Πέρας. 44 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ακολουθεί η επόμενη ψηφοφορία για το πρωτόκολλο για την ε, απάλληψη του παράνομου εμπορίου σε καπνικά προϊόντα και εν προκειμένου η είναι η κυρία, Μαρτίνα Άντερσον. Άρα, δεν έχουμε κατατεθειμένες τροπολογίες, μία μόνο τροπολογία, λέει ο πρόεδρος, ή μάλλον καμία, καμία. Άρα, τελική ψηφοφορία τότε. Με συγχωρείτε, είμαι και εγώ λίγο κουρασμένο. Μία λοιπόν ψηφοφορία τελική αρχίζει. Τέλο. Εγκρίνεται 47 ψήφοι υπέρ, μία κατά και δύο αποχέ. Συγχαρητήρια. Ακολουθεί ο νέος μορφότυπος για προξενικές θεωρήσεις και πρόκειται για την απόφαση να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Η συγκήτρια είναι η κυρία Σίλβια Ιβόν Κάουφμαν. Μοναδική ψηφοφορία για την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 46 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Θα διαβάσω τώρα τα ονόματα των προσώπων που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική ομάδα. Shadow Rapporteur Petri Sarvama, Shadow Rapporteur, for, sorry, for that was for the EPP, Shadow Rapporteur for the ECR, Timothy Kirkhope, Shadow Rapporteur for Aldi, Gerard Dupre, Shadow Rapporteur for GUI NGL, Costas Chrysigonis, um, Shadow Rapporteur for the Greens, Bodil Valero, and the Shadow Rapporteur for the FTD is Beatrix von Stork. Thank you, colleagues. We move on to... Ευχαριστώ πολύ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Προχωρώ στο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Ταξιδιού για επιστρέφοντες επικός τρίτων χωρών. Και έχουμε και εκεί διαπραγματεύσει κτλ. Πρόκειται για μια και μοναδική ψηφοφορία. Με συγχωρείτε μια στιγμή να μου δώσουν την λίστα ψηφοφορία. Colleagues, if you just pause for one second, I'm going to get my correct voting list. Είναι λοιπόν ε, εισηγητή ο κύριο Γιούση Χαλαάχο. Συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Έχουμε μία οριζόντια συμβαστική τροποποίηση του κειμένου. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 20. Συνάδελφοι, έπρεπε ήδη από την αρχή να έχω αναφέρει ότι η κυρία Βερζιά ζήτησε προφορική τροπολογία στην τροπολογία 20 πριν το ε, convention να έχουμε τη λέξη European, Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ε, νομίζω ότι είναι αυτονόητη, αλλά δεν ξέρω αν η κυρία Βερζιά θέλει να ε, δώσει κάποια εξήγηση ή όχι. Αν συμφωνείτε όλοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην τροπολογία και ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 20. We already voted Amendment 20. Την ψηφίσαμε ήδη. Right, amendment 20. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, τροπολογία 20, αρχή της ψηφοφορίας. Amendment 20, colleagues. Τροπολογία 20. Κυρία Βερζιά, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να ζητήσω το λόγο για να διευκρινίσω ότι έχει διατυπωθεί λάθος η τροπολογία αυτή που περιλαμβάνεται λάθος στη συμβιβαστική. Το θέμα είναι ο σεβασμός της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξαφνικά βλέπω όλα τα κόκκινα φωτάκια που ανάβουν και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί όλοι να είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Yeah, θα ψηφίσουμε την ε, τροπολογία 20, 30, συγγνώμη, θα φτάσουμε εκεί, αλλά σας ρώτησα αν θέλατε να πάρετε το λόγο. Λοιπόν, 20 ε, και 21. Μπορούμε παρακαλώ να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 21. Λοιπόν, λήξη της τροπολογίας για την τροπολογία 20. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21, αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12, αρχή της ψηφοφορίας. Τροπολογία 75, όχι 74, διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 74, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14, αρχή της ψηφοφορίας. Κατά τμήματα, το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 80, αρχή της ψηφοφορίας. 8-0, 80. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 87, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15, αρχή της ψηφοφορίας. Τροπολογία 15, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 91, αρχή της ψηφορίας. 91. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 90. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 92. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. 94. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 19. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 από τις αιτιολογικές σκέψεις. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 22, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Η κυρία Βερζιά ζήτησε προφορική τροπολογία μας εξήγησε περί τίνος πρόκειται, αρχή της ψηφοφορίας. Ε, ευγενικά το λέω. Πολύ καλά το εξηγήσατε. Εγώ τα μπέρδεψα τα πράγματα. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία ε, συμβαστική 7, κατά τμήματα, το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 42. Όχι, καταπίπτει. Τροπολογία 5, κατά τμήματα, το πρώτο, το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Αρχή της ψηφοφορίας. Το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πενήντα δύο, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 53. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Ε, τροπολογία 7, το πρώτο τμήμα. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57. Κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 59. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 63. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Αρχή της ψηφοφορίας. Συγγνώμη, κατά τμήματα, το πρώτο τμήμα. Αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 64, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 65. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 68 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12, το πρώτο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 39 υπέρ, 9 κατά, 2 αποχές. Και επίσης ε, ψηφίζουμε την απόφαση για την ενέργεια των διαπραγματεύσεων ε, με απόλυτη πλειοψηφία αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 35 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια. Check 11? The, the last one, yes. Content and order. Yeah. We're taking one more vote, colleagues. Um... No, I... Άλλη μία ψηφοφορία έχουμε. Α, όχι, ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η ώρα της ψηφοφορίας. We have one more, colleagues, we have one more item of business. we... Άλλο ένα θέμα έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Um, το τελευταίο σημείο είναι το σημείο 11. Δεν ψηφίζουμε, είναι θέμα προσυζήτηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, παρακαλώ να σεβαστείτε τον επόμενο εισηγητή. Σας παρακαλώ να κάνετε λίγη ησυχία για ένα τελικό σύστημα ΦΠΑ και για καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η συγητής... Είναι ο Χουάν Φερνάντες Λόπες Αγγιλάρ. Είναι έτοιμος να παρουσιάσει λοιπόν την πρώτη του πρόταση για την έκθεση πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση του ΦΠΑ. Χουάν Φερνάντο, έχει το λόγο. Κοιτάξτε, είναι το τελευταίο σημείο. Παρακαλώ όσοι θέλουν να φύγουν να το κάνουν με ησυχία. Ο Χουάν Φερνάντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Α, συνειδητοποιώ ότι είμαστε λίγο εξαντλημένοι μετά από μια μακρά ψηφοφορία. Αυτό είναι φυσιολογικό αλλά θα χρειαστούμε πολύ λίγα λεπτά για να μοιραστούμε με όσους αντέξουν κάποια σχόλια για το θέμα που έχουμε μπροστά μας, ένα σημαντικό νομίζω θέμα, ε, σχετικά με ποινικέ κυρώσεις, ε, σχετικά με την οδηγία ΠΥΦ την οδηγία δηλαδή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέτρα ποινικού χαρακτήρα. Η εργασία είναι σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε δουλειά ακόμα. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζετε ότι είναι κομβικό σημείο ε, της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών έτσι ώστε να τους διαβεβαιώσει ότι τα χρήματά τους θα χρησιμοποιηθούν με τον σωστό τρόπο. Συνειδητοποιώ ότι η εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειούται τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε πλέον το μέσο ανάκτησης τμήματος της απολεστής σας εμπιστοσύνης. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς της Europol, 40 με 60 εκατομμύρια σε επίπεδο ΦΠΑ απώλειες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης του οργανωμένου εγκλήματος και το 2% αυτών των ομάδων καλύπτει και προκαλεί το 80% της απάτης της λεγόμενης καρουσέλ. Το γαϊτανάκι θα λέγαμε είναι κάτι το οποίο επιτρέπει να υπάρξει φοροδιαφυγή σε ΦΠΑ σε πολύ ψηλά επίπεδα. Είναι ε, λυπηρή η κατάσταση λόγω και της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την οικονομία μας και την ανάπτυξή της και την ανάκαμψή της. Οι διαπραγματεύσει Συμβουλίου Κοινοβουλίου για την οδηγία αυτή, η λεγόμενη ΠΙΦ, προς το παρόν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένας βασικούς από τους λόγους είναι η συμπερίληψη της οδηγίας αυτής ή μάλλον στο εσωτερικό της οδηγίας αυτής των σημείων που θέτει το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν έχει αποδεχθεί ακόμα παρά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, την απόφαση Ταρίκο και άλλες τουλάχιστον οκτώ αποφάσεις ε, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που εκδόθηκαν το 2015 και που ξεκαθαρίζουν οι αποφάσεις αυτές ότι το ΦΠΑ θα πρέπει να θεωρηθεί πόρος χρηματοδοτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα κάνει μία έκθεση πρωτοβουλία λοιπόν για ένα τελικό τέτοιο σύστημα που θα επιτρέψει και την καταπολέμηση της απάτης. Οι συνεργαζόμενες επιτροπές ε, είναι η ΛΥΜΠΕ και η ΦΡΟΝΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού. Για τα θέματα που άπτονται των δικών μας λοιπόν αρμοδιοτήτων, εγώ θεωρώ ε, ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε την, να στηρίξουμε την ε, γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ με τα σημεία που ακολουθούν. Συμπερίληψη της, ε, του ΦΠΑ στην οδηγία ΠΙΦ, προώθηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ανεξάρτητης εισαγγελίας της ΕΠΟ, έτσι ώστε να παραπέμπονται στα δικαστήρια αυτοί οι οποίοι διαπράττουν εγκληματικές ενέργειες σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΙΦ, της οδηγίας ΠΙΦ. Νομίζω ότι η οδηγία αυτή είναι κάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα δημιουργήσει την δυνατότητα για τον Ευρωπαίο εισαγγελέα να αναλάβει ε, τον ρόλο του και να αυξήσει τις αρμοδιότητες του. Δυστυχώς όμως η λογική αυτή αμφισβητείται από χώρες στο Συμβούλιο και εγώ είμαι πεπισμένος ότι η αδίποτε ασθενέστερη λύση θα είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει απώλεια οικονομική για τον προϋπολογισμό μας. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση του αναδιόμενου λαϊκισμού και ευρωσκεπτικισμού είναι σε σχέση με την διαχείριση του δημοσίου χρήματος να είμαστε αποτελεσματικοί. Απαιτείται λοιπόν να αναλάβουμε δράσεις το ταχύτερο δυνατόν και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω να συνεχίσουμε την πίεση προς το Συμβούλιο έτσι ώστε να σταματήσει να κολλησιεργεί γύρω από το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Εγώ συζήτησα το θέμα αυτό με το Συμβούλιο επανειλημμένα. Το συζήτησα και με την Ολλανδική Προεδρία και με την επόμενη Προεδρία. Ε, έχει φτάσει η στιγμή να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια αυτή και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων πάνω σε αυτό. Στη γνωμοδότησή μας λοιπόν στην έκθεση της ΕΚΟΝ για το νομικό καθεστώς του ΦΥΠΙΑ. Πρέπει επιτέλους να είμαστε αποτελεσματικοί και να ξεπεράσουμε την αδράνεια στην οποία έχουμε περιπέσει στα πλαίσια της οδηγίας Πυφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάνω. Υπάρχουν κάποιοι παρόντες σκιώδεις. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπόνι για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκπροσωπώ τον Τόμα Στεχόφσκι και το Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ τον Χουάν Φενάντο Λόπες Αγουιράρ για την θαυμάσια οργάνωση της εργασίας για να φτιαχτεί ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και να μπορέσει να καταπολεμηθεί απάτη, η απάτη ε, ΦΠΑ, πάντοτε υπήρξε προτεραιότητα. Χρειάζεται ενίσχυση του Eurofix, συντονισμός των ενεργειών των εθνικών αρχών αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όπως Ευρωπόλ, Eurojust, Olaf κλπ. για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έκτημα και το ξέπλυμα του χρήματος. Η πολιτική μας ομάδα αποδίδει μεγάλη αξία στη, στο σχέδιο εκθέσεως. Γιατί και η οδηγία και το APPO είναι σημαντικά πράγματα και δεν ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Θα θέλαμε λοιπόν να εγκριθεί σύντομα και αυτό ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος Μωράης. Άλλος κανείς παρακαλώ επιθυμεί να λάβει το λόγο. Όχι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Ε, η ΠΠΟ σημειώνει διερμηνία στην Ευρωπαϊκή Αγγελία. Μέχρι τις 2 Ιουνίου λοιπόν κατάσταση τροπολογιών 12η μεσημβρινή. Ευχαριστώ για την παρουσία του θέματος. Λυπούμε που ήταν κάπως ε, θορυβόδης η ατμόσφαιρα πριν να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και ιδίως εσάς που μείνατε μέχρι τέλους άλλα θέματα, υπό τα διάφορα. Όχι. Ωραία. Υπό την αίρεση της εγκρίσεως η επόμενη συνάντηση θα είναι την ημερομηνία που προβλέπετε και τη βλέπετε στα έγγραφα. 13 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ.